Ευχαριστώ αγαπητέ συνάδελφοι. Δυστυχώ δεν ήταν διαδικαστική η παρέμβασή σα. Δεν έχετε το δικαίωμα να ρωτήσετε την Κομισιόν μέσα στην κανονική διαδικασία. Έχουμε έξι ψηφίσματα τα οποία ψηφίζονται τώρα. Το χθεσινό, τα χθεσινά πρακτικά και τα κείμενα τα οποία έχουν εγκριθεί είναι ήδη δημοσιευμένα. Υπάρχουν κάποιες αντιρρήσεις σε σχέση με αυτά τα πρακτικά. Εάν όχι. Εγκρίνονται. Και τώρα περνάμε στην ψηφοφορία. Ψηφίζουμε καταρχάς το κοινό ψήφισμα για έξι προτάσεις ψηφισμάτων για τη Μαλαισία. Κύριε Πρέντα. Κύριε Πρόεδρε. Πρόεδρε. Θα ήθελα να ζητήσω εξ ονόματος πολιτικής μου ομάδος όταν γίνει η ψηφοφορία για τους πρόσφυγες από την Ερυθρέα εμείς να κάνουμε ονομαστική ψηφοφορία για την πρόταση του ΕΛΚ και να πούμε όχι εμείς στο άλλο κείμενο. Ο πρόεδρο. ακούσατε τη ζήτηση ο συνάδελφο. Αν δεν υπάρχουν αντιρρήσει θα ακολουθήσουμε την πρότασή του. Δεν βλέπω αντιρρήσει. Ψηφίζουμε τώρα το κοινό ψήφισμα για την Μαλαισία. Τροπολογία υπαριθμών 2. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Αιτιολογική σκέψη Z, G. Τροπολογία 1 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται η πρόταση ψηφίσματος στο σύνολό της υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Και τώρα ψηφίζουμε έξι προτάσεις ψηφισμάτων για την Ουγγάντα Πρώτα το κοινό ψήφισμα έχει ζητηθεί χωριστή ψηφοφορία για την υπαριθμόν 7 παράγραφο υπέρ κατά το σύνολο του ψηφίσματος ονομαστική ψηφοφορία άρχεται η ψηφοφορία Haben alle Kollegen abgestimmt? όλοι. Πέρας της ψηφοφορίας εγκρίνεται το ψήφισμα. Και τώρα προχωρώ για την ψηφοφορία επί έξι προτάσεων ψηφίσματος για τους ερυθρέους πρόσφυγες που κατούνται όμοιροι στο Σινά. Έχουμε καταρχάς το κοινό ψήφισμα, παράγραφος 5 του αρχικού κειμένου, σε δύο τμήματα, πρώτο τμήμα υπέρ, κατά αποχές. Απορρίπτεται το δεύτερο τμήμα παρακαλώ. Βεβαίω, ζητείτε επαλήθευση, άρχεται η ηλεκτρονική επαλήθευση. Εψήφισαν όλοι. Πέρα τη ψηφοφορία. Απορρίπτεται. Καταπίπτει έτσι και το δεύτερο τμήμα και περνάω στην παράγραφη αριθμών 9 του αρχικού κειμένου υπέρ. Κατά. Επαληθεύουμε και πάλι ηλεκτρονικά παράγραφος 9. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψήφισαν όλοι. 25 υπέρ 37 κατά απορρίπτεται και τώρα ψηφίζουμε το ε, τροποποιημένο ψήφισμα υπέρ κατά Ονομαστική ψηφοφορία δεν έχουμε τώρα, έτσι, δεν είναι ονομαστική ψηφοφορία. Ο κύριος Πρέτα εξήγησε ότι ήθελε την ονομαστική ψηφοφορία όχι για το κοινό ψήφισμα, αλλά μόνο για, το, για την πρόταση για ονομαστική ψηφοφορία, για την πρόταση του ΕΛΚ. Αλλά αν θέλετε, αφού αμφισβητείτε και το αποτέλεσμα, ας κάνουμε ηλεκτρονική επαλήθευση. Εψήφισαν οι πάντες πέρα στις προφορίες. Απορρίπτεται. 31 υπέρ, 31 κατά. Τώρα ψηφίζουμε τα επιμέρους ψηφίσματα. Καταρχάς των φιλελευθέρων Β7, 7, 12, 2010. Υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. Σοσιαλιστές και Δημοκράτες 7, 7, 15, 2, 10. είναι υπέρ αυτού του ψηφίσματος. Κατά. Απορρίπτεται. ECR, ε Ευρώπη των Στηριωτικών και των Μεταρρυθμιστών, με, μάλλον όχι, κάνουμε παλήθευση για το προηγούμενο ψήφισμα των Σοσιαλιστών Δημοκρατών. Άρχεται η ψηφοφορία, ηλεκτρονική επαλήθευση. Το Β7715 των σοσιαλιστών. εψήφισαν οι πάντε. Ολοκληρώνεται η ψηφοφορία. Απορρίπτεται. Και τώρα περνάμε στο 7719 του 210 των ECR με ηλεκτρονική επαλήθευση. Άρχεται η ψηφοφορία. Εψήφισαν οι πάντες. Πέραση ψηφοφορία. Απορρίπτεται. Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματο. Με προφορικέ τροπολογίε. Πριν από την πρώτη παράγραφο, προφορική τροπολογία του κυρίου Κασίνη. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Η τροπολογία αυτή έχει σαν στόχο να είναι πιο ξεκάθαρη καταδίκη μας ως προς τη συμπεριφορά της Αιγύπτου. Όχι μόνο να σημειώσουμε ότι κάτι κάνει η Αίγυπτος, αλλά να ζητήσουμε άμεση απελευθέρωση και παρέμβαση της Αιγύπτου, άμεση απελευθέρωση αυτών των ομήρων. Και γι' αυτό θα πρέπει να μην επιβάλλονται ε, μέτρα δίωξης εις βάρος αυτών των ε, ομήρων που προσπαθούν να περάσουν τα σύνορα, να μην ασκείται δηλαδή βία εις βάρος τους, αλλά να διευκολυνθούν ε, ώστε να, και πάνω απ' όλα να απελευθερωθούν αυτοί οι όμοιροι. Το κείμενο λοιπόν λέει ότι θα πρέπει οι Αιγυπτιακές αρχές να βοηθήσουν στην απελευθέρωση των ομήρων αποφεύγοντας την χρήση ακόμη και θανάσιμης δύναμης εις βάρος των ανθρώπων αυτών όταν θέλουν να περάσουν τα σύνορα, σεβόμενες την σωματική και ψυχολογική του υγεία και εξασφαλίζοντα του τη δυνατότητα πρόσβαση στην υπατιαρμοστία των Ηνωμένων Αθηνών για του πρόσφυγες και αντίστροφα. Το κείμενο αυτό θα μπει πριν από την παραγραφό. Ένα. Υπάρχουν αντιρρήσει κατά της προφορικής τροπολογίας. Όχι. Ψηφίζουμε λοιπόν. Προφορική τροπολογία ψήφι υπέρ. Κατά. απόχε Απεφε, ούτω ενεκρίθη. Άλλη μια προφορική τροπολογία. Πριν από την παράγραφο 7 του κυρίου Σασόλη. Κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, ζητώ το ψήφισμα που δεν απέχω τόσο πολύ από το κείμενό του να προσθεθεί μια παράγραφος που μου είναι ιδιαίτερα προσφυλής που αφορά το σημείο 9 του κοινού ψηφίσματος. Το διαβάζω καλούμε τα κρατημένα να αντιμετωπίσουν την ανθρωπιστική κρίση μέσω της εθελοντική επανεγκατέστασης στην Ευρωπαϊκή Ένωση όλων των ζητώντων των ετούντων ασύλου στην κρίση και ζητά την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να συντονίσει αυτή τη διαδικασία με του πόρου του Ευρωπαϊκού Ταμείου Πρόσφυγων. Ευχαριστώ. Κύριε Κασίνη, χωρίς μικρόφωνο ο Θα ήθελα σαν ερώτημα να διευκρινίσετε η παρέμβαση η οποία αναφέρεται σε αυτούς που ζητούν το δικαίωμα ασύλου. Σε αυτούς που έχουν το δικαίωμα ασύλου. Είναι επικίνδυνο το να πούμε σε αυτούς που ζητούν το δικαίωμα ασύλου. Πρέπει να πούμε σε αυτούς που έχουν το δικαίωμα ασύλου. Εγώ θα ήθελα να ζητήσω από τον εισηγητή να πει όχι αυτοί οι οποίοι ζητούν άσυλο, αλλά αυτοί που έχουν το δικαίωμα σε άσυλο. Ζητούμε από την Επιτροπή. Όχι, όχι, όχι, όχι, λέει ο πρόεδρο. Κύριε Σασόλη, όχι. Κύριε Σασόλη. Δεν μπορούμε να μπούμε τώρα σε νέα συζήτηση. Σας έχει κάνει μία, έχει αντιταχθεί στο θέμα αυτό. Υπάρχουν αντιρρήσει διαδικαστικά για την ε, προφορική αυτή τροποποίηση. Όχι, την ψηφίζουμε. Ψήφι υπέρ. Δεν ήταν 40 οι οποίοι σηκώθηκαν, θα ήταν πολύ δύσκολο να βρεθούν 40 βουλευτές. Ψηφίζουμε αυτήν λοιπόν την ε, προφορική τροπολογία. δεν είσαστε αρκετοί. Λοιπόν, ψηφίζουμε αυτή την τροπολογία επομένω. Ψήφι υπέρ την ε, τροπολογία του κ. Σασόλη μετά την παράγραφο 7. Κατά. Αποχές. Έχει απορριφθεί. Θέλετε να ελέγξουμε. Να ελέγξουμε. Άρχεται η, η ψηφοφορία ελέγχου. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Απορρίπτω. Τελική ψηφοφορία λοιπόν για το κείμενο του ΕΛΚ. Ηλεκτρονικά παρακαλώ. Άρχεται η ψηφοφορία. Ονομαστικά μάλιστα. Άρχεται ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Ενεκρίθη το ψήφισμα αυτό με 36, 14 και 10 αποχές. Εκπίπτουν τα υπόλοιπα ψηφίσματα επομένω. Εκ του Συμβουλίου έχω πάρει την θέση για την πρώτη ανάγνωση ορισμένων νομοθετημάτων τα οποία θα δημοσιευτούν στα πρακτικά της ε, τρέχουσας συνεδρίασης. Υπάρχει προθεσμία τριών μηνών το Κοινοβούλιο να δώσει τη γνωμοδότησή του να σταθμίσει στη θέση του από τις 17 Δεκεμβρίου 2010. Αναφέρονται λοιπόν στα πρακτικά οι τρεις αυτές προτάσεις του Συμβουλίου. Τα πρακτικά αυτής της συνεδρίασης θα εγκριθούν στην επόμενη συνεδρία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.